Allow me Επιτρέψτε μας να αρχίσουμε το δεύτερο τμήμα της σημερινής μας συνεδρίασης, της κανονικής μας δηλαδή συνεδρίασης. Καταρχήν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. έχουν αντιρρήσεις. Όχι, εγκρίνεται. Η διερμηνία είναι στις γλώσσες των πλήρων μελών της Υποεπιτροπής. Και υπάρχει και αναμετάδοση. Πρώτο θέμα μας είναι το θέμα του κυρίου Πάσκου, η έκθεση του κυρίου Πάσκου για τη στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας μετά από την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Είναι πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Το έγγραφο έργαση του κυρίου Πάσκου διανεμήθηκε στα μέλη. Και τώρα του δίνω το λόγο. Ιωάν Μίρτσα Πάσκου. Σας κατευχαριστώ. Η παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία άλλαξε πλήρως τη στρατηγική και στρατιωτική κατάσταση γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είχε επιπτώσεις σε πολλές κατευθύνσεις. Πρώτον, αν η Ρωσία κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι πλησιάζει τη Ρωσία, τώρα η Ρωσία προσέγγισε το ΝΑΤΟ και σε μήκος εκατοντάδων χιλιόμετρων δεύτερον. Τα, συστήματα, τα πυραυλικά συστήματα που μπορούν να εγκατασταθούν και εκτός πλέον της Σεβαστούπολης αλλά σε ολόκληρη πια την, την ε, Κρυμαία καθιστούν ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη ευάλωτη. και την θέτουν σε κατάσταση υπό Και αυτό έχει σημασία και στρατηγικός και τακτικός στρατηγικά μέχρι και για την ε, Μέση Ανατολή και τακτικά και για την υπερθενιστερία. Τώρα η Ρωσία έχει σύνορα με τη Ρουμανία που είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Θαλάσσια σύνορα. και το άνοιγμα από την Οδυσσό στην Υπερνηστερία όπως ξέρετε η Οδυσσός ε, αφορά και την Μαριούπολη που είναι για την Αζωφική θάλασσα και για τη Ρωσία πολύ σημαντικό άνοιγμα και είναι απέναντι από την Οδυσσό. Επίσης αμυντικά η Ρωσία ενδυναμώθηκε από την προσάρτηση της Κρυμαίας γιατί κατέστησε την Αζωφική θάλασσα ρωσική θάλασσα και επίσης ενδυναμώνει στρατηγικά όλο το νότιο τμήμα της Ρωσίας από τη Μαύρη Θάλασσα. Η προσάρτηση έχει και άλλες επιπτώσεις και οικονομικές διότι υπάρχουν τα ουκρανικά κοιτάσματα αερίου και πετρελαίου που τα πήρε και αυτά η Ρωσία και η Ρουμανία είχε μερικά κοιτάσματα κοντά στα Ουκρανικά που τώρα έγιναν Ρωσικά και από την Κρυμαία η Ρωσία τώρα μπορεί να ελέγξει όλες τους διαδρόμους για το αέριο και το πετρέλαιο. Κάτι άλλο είναι η ναυτική ισορροπία στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας η Ρωσία έκανε μια πολύ ένα πολύ επιθετικό εξυγχρονισμό του στόλου της και η Τουρκία είχε αρχίσει να εφαρμόζει μια, ένα τέτοιο εξυγχρονισμό και τον σταμάτησε. Και τώρα οι αναλύσεις λένε ότι θα καθυστερήσει, θα έχει υπεροπλία η Ρωσία. Θα δούμε αν η Τουρκία μπορεί να αντιδράσει. Οι στρατιωτικές δομές επίσης. Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες στη Μαύρη Θάλασσα. Η μία λέγεται Black Sea που είναι μια ελάχιστη συνεργασία μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων εκεί για επιχειρήσεις διάσωσης κλπ. Και μια άλλη πρωτοβουλία τουρκική από το 2004 λέγεται Blue Harmony. Επίσης οι επιπτώσεις οι μελλοντικές ναυτικές επιπτώσεις δεν είναι ακόμη γνωστές. Γιατί δεν υπάρχουν δομές που να αναλάβουν τέτοιες μελέτες. Θα έλεγα ότι μακροπρόθεσμα η συνεργασία με τη Ρωσία είναι προτιμότερη από την ε, αντιπαράθεση, αλλά εντωμεταξύ ξέρετε ότι οι χώρες της περιοχής θέλουν μεγαλύτερη στρατιωτική μεγαλύτερο στρατιωτικό καθησυχασμό. Γιατί υπάρχει και η υπονόμευση που δεν την καλύπτει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Δεν προβλέπει την υπονόμευση, μόνο κλασικές επιθέσεις Αλλά όπως έκανε και το ΝΑΤΟ για τις κυβερνοεπιθέσεις πρέπει ίσως να διευρύνουμε τον ορισμό του τι είναι επίθεση. Και τώρα για να καταλήξω θα έλεγα ότι η Κρυμαία η Κρυμαία λέγω ε, είναι περίπτωση παραβίασης των κανόνων καλής γειτονίας και καλής συμπεριφοράς και δεοντολογίας Ξέρετε το πρωτόκολλο της Βουδαπέστης αφορά συγκεκριμένα την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Το επιχείρημα της Ρωσίας ότι η Κρυμαία κάποτε ανήκε στη Ρωσία είναι, δεν ισχύει γιατί πολλές χώρες έχουν περιφέρειες που τώρα δεν είναι δικές τους. Και αν αρχίσουν όλοι να χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα δεν θα μείνει τίποτα στην Ευρώπη. Uh, για ιστορικούς λόγους. Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Έχουμε τώρα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν την δυτική στάση, δηλαδή μία αναγνώριση της προσάρτησης που θα παραμείνει όσο χρειαστεί και κυρώσεις για ό,τι αφορά την Κρυμαία. Επίσης θα έλεγα καταληκτικά ότι δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα. Από τη μία θα συνεχιστεί η έρευνα και η μεταφορά αερίου και πετρελαίου, αυτό είναι το θετικό. Από την άλλη όμως το αρνητικό είναι ότι θα γίνει μάλλον ε, ένας αγώνας στρατιωτικών ναυτικών δηλαδή εξοπλισμών και ό,τι κερδίσει κανείς από εκεί θα αντισταθμιστεί από τις απώλειες στρατιωτικά. Η Ένωση είναι παρούσα εκεί αλλά δεν θέλησε να ξεπεράσει τα όρια αυτής της συνέργειας πράγμα που είναι απλώς ένα άλοθη για να μπορούν να πούνε Εντάξει, το λύσαμε. Αυτή ήταν η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν βλέπω κανένα θάρρος σε αυτήν τη στάση για να βελτιωθεί η συνέργεια και να γίνει στρατηγική που τη ζήτησαν άλλες εκθέσεις από το 11 ήδη. can Δεν ξέρω αν η Ένωση θα προχωρήσει προς την κατάρτιση στρατηγικής, αλλά είναι θέμα όπου πρέπει να συνεργαστεί το ΝΑΤΟ με την Ένωση. Γιατί οι αλλαγές αφορούν και τις δύο οργανώσεις. Ευχαριστώ. Rest my Thank you, Mr. Pascu, for this. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πάσκου για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρέμβαση. Πρόκειται βέβαια για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την έκθεση. Έτσι κάνουμε συνήθως. Και τώρα πρέπει οι σκιώδεις εισηγητές να πάρουν το λόγο. Ο ε. κύριος Καπριέλ Λαντσμπέργκης, εκ μέρους του ΕΛΚ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έγγραφο εργασίας. Νομίζω ότι μας ε, έδωσε τις αντρές γραμμές της εκθεσής του πολύ ξεκάθαρα. Να πω τρία πράγματα. Πρώτον, από ό,τι βλέπουμε, κατάσταση στην Κρυμαία σήμερα νομίζω ότι είναι απλά και μόνο η αρχή μιας αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης. Κάθε εβδομάδα παίρνουμε αναφορές για νέα σκάφη ε, πλοία και πυρηνική ίσως ε, ικανότητα. Και αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να αλλάξει ίσως και τη στρατηγική κατάσταση συνολικά σε όλη την Λεκανική. Άρα μία λύση θα μπορούσε να είναι να συζητήσουμε αλλάζει η κατάσταση, την κατάσταση αυξημένη στρατιωτικοποίηση έχουμε status quo. Τι περιμένουμε για το μέλλον. Δεύτερον, το αναφέρατε και εσείς εν μέρη και είναι και στο έγγραφο εργασίας. Μιλώ για ένα είδος υβριδικού πολέμου, μια υβριδική ε, απειλή. Ενέργεια, πληροφορίες, κυβερνοχώρος. Πώς μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από την ε, κατάσταση στην Ουκρανία. Για τις ε, χώρες που είναι άμεσα ε, για την σας προς την λεκάνη του Ευξενού Πόντου, της Μαύρης Θάλασσας και γενικότερα. Τρίτον, ένα θέμα το οποίο νομίζω δεν μπορεί να τεθεί μόνο σε αυτή τη συζήτηση, αλλά θα μπορούσε να τεθεί και αλλού σε άλλα βήματα συζήτηση. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την περιοχή. Διότι όποτε συζητάμε για την ανατολική εταιρική σχέση, λέμε ότι πρέπει να έχουμε μια ατομική προσέγγιση, εξατομικευμένη προς κάθε χώρα. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για τις ε, χώρες ε, της συνεργασία. συνεργασίας. Θα μπορούσαμε να δούμε ίσως τη συμφωνία σύνδεσης. Έχουμε τώρα τρεις τέτοιες συμφωνίες, έχουν υπογραφεί. Και σε ένα απόσπασμά τους λέει αυξημένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Ίσως εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο φιλοδοξίες για το μέλλον, για να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία με τις χώρες της Λεκάνης. Γιατί βλέπουμε σε κάποιες να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και σε άλλες όχι. Δηλαδή κάποιες να δηλώνουν ενδιαφέρον για μεγαλύτερη συνεργασία και στον τομέα αυτό που σας ανέφερα και να μπορούμε εκεί να προχωρήσουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάντω για μία ακόμη φορά για το έγγραφο εργασία και είμαι βέβαιο ότι θα έχουμε καλή συνεργασία και στο μέλλον. Thank you. Uh... Ευχαριστώ πολύ. Ο σκιώδη της ομάδας ECR. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει, το έκανε ο προλαλής σας. Ε, καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί παρουσίασε με απόλυτη σαφήνεια το θέμα με το οποίο ε, πρέπει να ασχοληθούμε και τα έκανε όλα αυτά με απόλυτη σαφήνεια. Η κατάσταση στην Κρυμαία είναι πάρα πολύ σημαντική και λόγω των επιδιώξεων της Ρωσίας και ε, ευρύτερα λόγω των ε, προβλημάτων που προκύπτουν. Η δική μας η πολιτική δεν ε, είναι στο ύψος των καταστάσεων. Ο κύριος Πασκού το είπε και το έχει πει επανειλημμένα και η κυρία Μογκερίνη. Η κυρώσεις, οι οικονομικές κυρώσεις εφαρμόζονται και είναι το βασικό μας εργαλείο στον αγώνα αντιμετώπισης ε, αυτών των απειλών. Και όλα αυτά έχουν σχέση με την αποκλιμάκωση της ε, έντασης. Ε, κατ' ουσίαν δεν πρόκειται για την προσάρτηση της Κρυμαίας γιατί η προσάρτηση της Κρυμαίας είναι πλέον μια κατάσταση που αλλάζει τα πάντα και τα θέματα δεν περιορίζονται σε λεκτικό επίπεδο. Καλούμεθα όμως ε, να βρούμε μια πολιτική λύση και εδώ πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, εφάνταστοι όσον αφορά την απάντησή μας προς τη Ρωσία, μια απάντηση που να μην είναι μακριά από την πραγματικότητα. Τίθεται το ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει το μνημόνιο της Βουδαπέστης, το οποίο όμως πλέον δεν ισχύει. Και ακούμε τις προσδοκίες της Ρωσίας σε σχέση με το μνημόνιο της Βουδαπέστης. Ε, τότε όμως επρόκειτο για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Και το μνημόνιο της Βουδαπέστης ε, υποτίθεται ότι θα αντικαθίστατο από μια νέα συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και τις ε, όμορες χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Πάντως δεν μπορούμε να απεκδιώμεθα των ε, ευθυνών μας που είναι καταχωρημένες στην συμφωνία στο μνημόνιο της Βουδαπέστης η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι μια συμμετρική αντίδραση. Η Ρωσία άλλαξε το συσχετισμό δυνάμεων στην περιοχή και ως εκ τούτου και η Δύση θα πρέπει να αλλάξει την κατάσταση ε, σε σχέση με τις ε, βαλτικές χώρες οι οποίες δέχονται απειλή από τη Ρωσία. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι στην τελευταία συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ ετέθη το θέμα. Ε, σωστά ήταν όλα αυτά που ελέγχθησαν, αλλά βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον ε, προβάλλουν σωστά και κατά πόσον είναι η, η σωστή μας αντίδραση. Κάτι άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να εντείνουμε τη συνεργασία μας με τη Γεωργία. η Ρωσία λίγους μήνες ε, μετά την προσάρτηση της ε, Ρωσίας έκανε και άλλα βήματα σε σχέση με την απόσχηση της ε, Απχαζίας. Και κάτι άλλο που νομίζω θα τεθεί και πάλι επιτάπητος. Πρόκειται για τις αντιδράσεις μας και πρέπει να δείξουμε ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο σε λεκτικές διαμαρτυρίες όσον αφορά την προσάρτηση της Κρυμαίας, αλλά θα αντιδράσουμε για να διεκδικήσουμε μια ισορροπία. Και η τελευταία μου παρατήρηση. Νομίζω ότι αυτά που είπε ο κύριος Πάσκου είναι χρήσιμα και χρήσιμη είναι επίσης και η ειλικρίνεια με την οποία αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση. Δηλαδή, τα θαλάσσια σύνορα με τη Ρωσία. Αυτά έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια. Και θέλω να πω ότι τα προβλήματα που ακούμε να υπάρχουν και που θίγονται και στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές, αυτά δεν είναι προβλήματα που απορρέουν από ιστορικές συγκρούσεις. Έχω κατά νου τις χώρες Βαλτικής και τις σχέσεις τους με τη Ρωσία, αλλά δεν είναι αυτό το διακύβευμα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να παραμένει αξιοπιστία, να διασφαλίζεται η ασφάλεια των κρατών μας και να έχουμε μια σωστή αντίδραση, να μην περιοριζόμαστε μόνο σε διπλωματικές ε, διαμαρτυρίες. Το θέμα είναι να αναγνωρίζουμε την ε, έκταση του προβλήματος. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που είπατε εκ μέρους ε, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών και επιτρέψτε μου να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Επόμενος ομιλητής. Ερνάν, ε, από άλλη, συγγνώμη. Η Κρυμαία για μένα είναι από το τμήμα της Ουκρανίας. Είναι σαφές, ε, είναι γνωστό ε, και υπάρχουν συνθήκες που επέγραψε η Ρωσία όταν ανεξαρτητοποιήθηκε η Ουκρανία και εκεί εγγυόταν και την ασφάλεια, τα σύνορα και την αδαφική ακαιρεότητα. Αυτό όμως έπαψε να ισχύει μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας Σα παρακαλώ, σας παρακαλώ. Πρέπει να έχουμε επίγνωση των λόγων που εξτομίζουμε. Σίγουρα η εισβολή και η προσάρτηση στην Κρυμαία είναι παράνομη και αντιβαίνει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Το ίδιο όμως ισχύει και με την ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου που παραβίασε το χάρτη του Ελσίνκη. Πρέπει να λέγονται οι αλήθειες, ε, γιατί για πραγματικότητες άλλων λέμε ότι είναι ψέματα. Και άλλο παράδειγμα έχουμε την ε, ε, Ελλάδα, την ε, Αρμανία, τη Σλοβακία και κάποιες άλλες χώρες. Στην αρχαιότητα μπορούσε οποιοδήποτε να διεκδικεί κυριαρχικά δικαιώματα στο εσκούδο του βασιλιά της Ισπανίας είναι και η φλάνδρα μέσα το Βέλγιο. Δεν πρόκειται αύριο όμως να πάμε εμείς να εισβάλλουμε στο Βέλγιο. Δεν μπορούμε λοιπόν να επικαλούμεθα την ιστορία. Όταν ήταν η Σοβιετική Ένωση ε, μόνη της ένα ειδηλικό βοσκότοπο, ο, Χρουτσεφ, ε, ο Χρουτσόφ συγγνώμη, ε, χάρισε την Κρυμαία, που κατοικείται κατά πλουσία από Ρώσους. Μπορεί να μας αρέσει πραγματικά αυτή, όμως έτσι είναι τα πράγματα. Άρα ξεκινάμε με μια εικασία είχαμε την εισβολή της Πολωνίας από τον Χίτλερ. Αλλά είναι αυτό διαφορετικό και έχει να κάνει με τη δόξη μιας χώρας με σύνορα που δεν αντιστοιχούν στις δημογραφικές πραγματικότητες. Πρέπει όμως να τα σεβαστούμε για να μην υπάρχει χάος. Και θυμίζω πάλι το κοσφοπέδιο. Η Ρωσία λέει ότι μπορεί να είναι κουτί, κουτί που θα ανοίξει ε, ασκό του αιώλου. Μόνο Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρος και άλλες δύο χώρες, δεν θυμάμαι ποιες, τα κατά. Μπορεί να μην μας αρέσει λοιπόν, αλλά πρόκειται για αντίστοιχη περίπτωση. Δεύτερο, σαν ε, η Μαύρη Θάλασσα άλλαξε ε, κατάσταση, η ε, θέση μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας. Κάτι άλλαξε, αλλά δεν άλλαξε και τίποτα σημαντικό γιατί υπήρχε η, βάση, η ναυτική βάση της ε, Σεβαστόπολης που δεν άλλαξε. Ήταν μια ρωσική βάση σε ουκρανικό έδαφος, αλλά ε, ήταν μια μόνιμη στρατηγική βάση ρωσική. Και δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον. Άρα μην λέμε ότι άλλαξαν άρδιν τα πράγματα από στρατηγικής πλευράς το ότι έγινε ε, η θάλασσα ε, αυτή ρώσικη μπορούμε να το πούμε, αλλά ε, τα στενά του Κέρσφ που χωρίζουν την Κρυμαία από τη Χερσόνησο του Κουμπάν πάντοτε ελεγχόταν από τη Ρωσία. Επομένως αυτή η θάλασσα παραμένει, να είναι, παραμένει μια κλειστή, μια περίκλειστη θάλασσα που την ελέγχει η Ρωσία. Από τη μία ελέγχονται τα στενά του ΚΕΣ, αλλά υπάρχουν δύο όχθες που ελέγχονται πλέον και αυτό πρέπει να το λέμε. Η Ρωσία είναι στα σύνορα με τη Ρουμανία, με την υπερδνηστερία, θα φτάσει και ε, στα σύνορα με τη ε, Μολδαβία. Η υπερδνηστερία όμως δεν έχει έξοδο προς τη θάλασσα, δεν έχει πρόσβαση. Φυσικά αυτή η αυτονόμηση, η απόσχηση της υπερνηστερίας ε, είναι κάτι που με βρίσκει αντίθετο, αλλά ε, και για τη Μολδαβία πρέπει να μιλήσουμε. Έχουμε μια τεχνητή προσάρτηση. Η Μολδαβία ποτέ δεν ε, πέρασε από την επόμενη του ΝΙΕΤ. Αυτό έγινε με εσωτερικές συμφωνίες στην ε, τότε Σοβιετική Ένωση. Μιλάμε για κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε μια ηγεμονική χώρα που λέγεται Ρωσία στην Μαύρη Θάλασσα. Το ίδιο ηγεμονικά φέρονται στον κόλπο του Μεξικού ΙΠΑ και κανείς δεν λέει ότι τα στρατηγικά συμφέροντα των ΙΠΑ είναι προτεραιότητα ε, και ηγεμονικά. Ε, και αναφέρομαι, και με εξαίρεση ε, οποιαδήποτε χώρα στον κόλπο του Μεξικού, και αναφέρομαι στην Κούβα. Η πιο μικρή χώρα του κόσμου έχει τα ίδια κυριαρχικά δικαιώματα με τη Ρωσία, την Κίνα, τη ΣΥΠΑ. Είναι σαφές αυτό. Δεν αντιμετωπίζουμε όμως όλες αυτές τις χώρες με τον ίδιο τρόπο για το λόγο του κοινού στρατηγικού νου. Δεν άκουσα μια λέξη σε σχέση με ένα πάρα πολύ σημαντικό μέλος ε, του ΝΑΤΟ που είναι στην Μαρθάλασσα και λέγεται Τουρκία και που ελέγχει τα Δαρδανέλια και είναι ε, ο σωματικότερος και ο μόνος στρατηγικός πρωταγωνιστής του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά το, στόλο, το ρωσικό στόλο της Σεβαστόπουλης που πρέπει ε, με βάση τη συμφωνία της, στην Ελβετία που είχαν υπογραφεί να πέρασει από τα στένα των Δαρδανελίων και των αεροπλανοφόρων την πρόσβαση ε, μέσω αυτών των συμφωνιών που ρυθμίζεται ακόμη. Όταν λέμε λοιπόν ότι η Ρωσία ελέγχει και τη αγούς πετρελαίου, μα έχουν αλλάξει τα πράγματα γιατί το South Stream θα περνάει από συμμαχική χώρα, από τη Ρωσία, ε, την Τουρκία. Από την Τουρκία η οποία όμως έχει αυτή τη στιγμή δυσκολίες στις σχέσεις της με τη Εν Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα το συστήσουμε τώρα εδώ. Υπάρχει ένα, μια εμπλοκή στις σχέσεις. Εμένα δεν μου αρέσει ο Πούτιν ούτε η προσάρτηση της Κρυμαίας και είμαι κατά όλων αυτών. Είναι όμως γείτονα, ε, δεν μπορούμε να τον παραγνωρίσουμε. Η γεωγραφία είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε ιδεολογικό βολονταρισμό ή ηθικό κριτήριο και με τη Ρωσία πρέπει να συμβιώσουμε. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να ε, φτιάξουμε μια στρατηγική σκακέρα στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Υπάρχει στρατηγική πρόκληση, είναι στα χέρια όμως των ΗΠΑ. Άρα οποιαδήποτε ε, στρατηγική αντιπαράθεση για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη δυσκολίες σχέση μας με τη Ρωσία που θα καταλήξει στο να δώσουμε όλα τα ατού στους φίλους και συμμάχους μας τους Αμερικανούς που δεν έχουν όμως τα ίδια συμφέροντα με τα δικά μας, τα ευρωπαϊκά έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Εγώ πιστεύω ότι και με βάση τις αρχές τις οποίες πρεσβεύω πρέπει να κατέβουμε λίγο και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγητής από την ΚΟΕ. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τον κύριο Πάσκου και να τον ευχαριστήσω για τη δουλειά του και γιατί ήταν πάρα πολύ ειλικρινής. Αλλά διαβάζοντας αυτό το έγγραφο εργασίας κύριε Πάσκου, δίνεται η εντύπωση ότι στόχος σας είναι να παίξετε με το χώρο και το χρόνο. Μιλάμε για ένα τετελεσμένο γεγονός από το Μάρτιο του 2014. Άλλαξε σίγουρα το γεωστρατηγικό σκηνικό, αλλά θα πρέπει όπως και κατά το παρελθόν ε, να δούμε τι γινόταν και ε, πώς αντιδρούσαμε παλιότερα, σαν ε, να μην υπήρχε καμία παρουσία της Ρωσίας. Ίσως να μην μπήκαν το, στο ΝΑΤΟ η Ρουμανία και η Βουλγαρία και μετά και στην Ένωση. Κάνουμε σαν να μην γίνεται τίποτα σε αυτή την περίπτωση όπως κάναμε πριν. Όχι. Έρχεται πιο κοντά στο ΝΑΤΟ η Ρωσία. Μήπως ε, το αντίστροφο συμβαίνει εδώ και 20 χρόνια προσεγγίζει το ΝΑΤΟ Ρωσία. Επίσης μιλάει το έγγραφο για την προσάρτηση της Κρυμαία και λέει ότι αψηφά το διεθνέ δίκαιο η Ρωσία και τους ε, διεθνού κανόνε, συμπεριφορά μεταξύ κρατών. Για μια ακόμη φορά εμείς ουσιαστικά ε, προσπαθούμε να χάσουμε την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Μάλλον έχουμε πρόβλημα μνήμης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Ε, έχουμε ένα πρόβλημα στην Επιτροπή. Δεν ξέρω πώς είναι μια νέα παθογένεια που είναι μια υπόρους αμνησία. Γιατί ούτε ο βομβαρδισμός του ΝΑΤΟ στη ε, το 1999 που στήριξαν τρομοκρατικές οργανώσεις που δούσαν τοπ, ούτε την αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου που το αναγνώρισαν τα περισσότερα ε, κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ το 8 ούτε ε, την παράνομη ε, μετατόπιση εξουσίας στην Ουκρανία. Αυτά δεν τα αναφέρουμε. Ε, με, λυπά, λυπεί το γεγονός που στην Ευρώπη η πλειοψηφία θέλει πάνω απ' όλα ε, να στηρίξει τον διατλαντικό δεσμό, όπως τον αποκαλεί. Και το μόνο που ζητά είναι αυτή την πολύ αθράυστη κατάσταση στην Μαύρη Θάλασσα, να την επηρεάσει ώστε τελικά να κυριαρχήσουν τα συμφέροντα των ΙΠΑ. Εγώ απευθύνω έκκληση να σκεφτούμε τα συμφέροντα της Ευρωπής. Γιατί είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να σκεφτούμε και τα συμφέροντα των λαών μας, των χωρών μας. Την ειρήνη να σκεφτούμε. Γιατί πάει πιο πέρα το θέμα από τις ιδεολογίες. Πρέπει να επιλέξουμε. Ή θα λύσουμε τα προβλήματα με τους γείτονες ή θα συνεχίσουμε να επακούμε, όσο επαγορεύει μια μεγάλη δύναμη. που όμως αυτοί μας έχουν κατατάξει σε δεύτερη κατηγορία, για τη ΣΥΠΑ μιλώ. Από τη στιγμή που πιο πολλοί στρέφονται στον άξονα Ασία-Ειρηνικού από ό,τι στην Ευρώπη, οι ηγέτε αυτή τη χώρα θεωρούν ότι ο καλύτερο τρόπο να μα κρατάνε υπό έλεγχο είναι να διατηρούν ε, ξεχωριστά και σε αντιπαράθεση μεταξύ του Ευρώπη και Ρωσία. Είναι σαφέ. Ή θα ε, υποκείμεθα σε μία ξένη στρατηγική και θα την υπακούμε ή θα υπακούσουμε και θα ε, προσπίσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Άρα πρέπει να απορρίψουμε αυτές τις προτάσεις και την άποψη του κυρίου Πάσκου, αν θέλουμε να κάνουμε το δεύτερο φυσικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο εισηγητής τώρα των Πρασίνων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήταν ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μέχρι τώρα. Άκουσα τις απόψεις των συναδέλφων. Είχα την εντύπωση ότι η άποψη του κυρίου Πάσκου θα μας έβρισκε αντίθετους, ε, κυρίως ε, γιατί εμείς είμαστε υπέρ της ειρηνικής συμβίωσης ε, και όλων των άλλων ε, στόχων των πρασίνων. Όμως τώρα βλέπω ότι δεν είμαστε εμείς ε, αναγκασμένοι να προβάλλουμε τους δικούς μας στόχους. Άλλοι το λένε αυτό. Και εγώ διαφωνώ. Εγώ συμφωνώ σχεδόν με όλα που είπε ο εισηγητής και πραγματικά θα κάνω ό,τι μπορώ για να πείσω και τους υπόλοιπους πράσινους συναδέλφους μου. Ο συνάδελφος από την ΚΟΕ έθεσε το ερώτημα ποια είναι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και νομίζω επ' αυτού πρέπει να εστιάσουμε την, πολιτική, την προσοχή μας στην ε, ΚΕΠΑ. Νομίζω ότι το είπαμε ήδη ότι αν ε, είχαμε ε, ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις μας στην κοινή αμυντική πολιτική δεν θα υπήρχε σήμερα το πρόβλημα της Κρυμαίας γιατί κανένας δικτάτορας δεν θα είχε ποτέ τολμήσει να αντιμετωπίσει μια κοινή εξωτερική πολιτική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα στηριζόταν και από μια κοινή αμυντική πολιτική. Και κάτι τώρα για το ΝΑΤΟ. Αν δούμε λιγάκι το ΝΑΤΟ και αφαιρέσουμε από αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε τι μένει η Τουρκία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και δεν νομίζω ότι συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο να αφήσει το ΝΑΤΟ στα χέρια ε, της Τουρκίας και, της, ε, και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, νομίζω ότι και αυτοί αξίζει να τους στήριξουμε και να τους υπερασπιστούμε. Το μόνο επί το οποίο διαφωνώ με τον κύριο Πάσκου είναι το εξής, ότι η Μαύρη Θάλασσα ελέγχεται τώρα από τη Ρωσία και αυτό είναι ε, κάτι το καινούριο ελέγχθη. Πράγματι κάποια κομμάτια της ε, ελέγχονται από τη Ρωσία αλλά κάποιοι απόστρατοι ναυτικοί ε, των Ηνωμένων Πολιτειών λένε ότι δεν είναι μεγάλη απειλή γιατί πολύ γρήγορα πούμε, θα μπορούσαν να δεχθούν μια αποτελεσματική επίθεση από τους Ιταλούς αν θέλετε. Ο η ναυτική τους δύναμη δεν αποτελεί καν ανταγωνισμό για μας. Δεν είναι ανταγωνιστική προς εμάς. Βεβαίως αυτό πάλι δεν δικαιολογεί την ε, επίθεση και την προσάρτηση μιας ε, ξένης χώρας. Και φτάνω τώρα στο αγαπημένο μου θέμα. Γιατί δηλαδή και πάλι στο πλαίσιο της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, γιατί Σκεφτόμαστε να δώσουμε κάποια λύση και στο γαλλικό πρόβλημα των σκαφών που θα μπορούσαμε να τα τοποθετήσουμε στα Δαρδανέλια. Εκεί γίνεται λόγος μόνο για ε, τα αεροπλανοφόρα που δεν επιτρέπεται να διασχίσουν τα Δαρδανέλια, όχι όμως για τα ελικοπτοφόρα. Και αυτό θα είναι το πρόβλημα. Ο κύριος Γκάλα, ε, μισό λεπτό. Κοιτάξτε, ε, λέει ο κύριος Γκάλα, κανονικά δεν θα είχα ζητήσει το λόγο για δύο λόγους. Πρώτον, διότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Πάσκου και ο δεύτερος είναι γιατί συμφωνώ και με αυτά που είπε ο Σκιώδης εισηγητής μας. Εγώ πρέπει όμως να σας πω ότι παρόλα αυτά πραγματικά ε, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η άποψη των ε, δυτικοευρωπαϊκών κομμουνιστών που παρουσιάζουν λάθος συσχετισμούς σε αντίθεση με τους ε, πρώην κομμουνιστές της Ανατολικής Ευρώπης οι δυτικοευρωπαίοι ακόμα δεν έχουν ε, βιώσει ή την ε, ήττα τους δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο να έχουν εξουσία πάνω σε συνανθρώπους και γι' αυτό παραμένουν σε καθαρά ιδεολογικό επίπεδο. Δηλαδή σήμερα υπεραμείνονται ενός Μιλόσεβιτς ο οποίος ήταν κομμουνιστής, μετά έγινε εθνικιστής, μετά έγινε ρατσιστής στο Κωσυφοπέδιο και ήθελε εκεί να διαπράξει γενοκτονία. Και μετά από 10 χρόνια, γιατί το 89 άρχισε το τέλος αυτονομίας στο Κοσμοπέδιο και χρειάστηκαν 10 χρόνια με διαπραγματεύσεις και όλα τα συμπαρομαρτούντα για να πούμε ότι δεν μπορούμε αυτό να το δεχτούμε. Μετά λοιπόν από 10 χρόνια επενεύει το ΝΑΤΟ για να αποφύγει, να παρεμποδίσει τη γενοκτονία και να το συνδέει κανείς τώρα αυτό με την Κρυμαία δείχνει ότι έχει ιδεολογικές ιδεολειψίες και αυτό ήθελα να επισημάνω ότι επουδενή δεν μπορεί κανεί να συγκρίνει ούτε πολιτικά ούτε νομικά την κατάσταση στο Κοσμοπέδιο όπου έπρεπε να προστατευτούν εκατοντάδες άνθρωποι πώς να το συγκρίνει κανείς αυτό με την προσάρτηση της Κρυμαίας. Συγγνώμη, εδώ δεν προβλέπεται ελεύθερη συζήτηση. Λοιπόν, ο κύριος Τσάρλς Τάνοκ, ε, αν ε, δεν κάναμε λάθος. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Πάσκο για τη δουλειά του. Εγώ συμφωνώ νομικά ότι η κατάσταση του Κωσυφοπεδίου είναι προβληματική γιατί δίνει δικαιολογία στη Ρωσία αλλά ηθικά δεν υπάρχει καμία σύγκριση, καμία και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε εκείνον που το είπε ότι ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτά που κάνει ο Πούτιν στη Ρωσία και που λέει ότι η Κρυμαία ιστορικά ήταν ρωσική. Έτσι και το Καλέ και το Μπορντό ήταν αγγλικά ιστορικά. Τα ίδια θα πούμε η Κρυμαία Αυτά που βλέπουμε τώρα είναι ότι δημιουργούνται αχυράνθρωποι και αχυροκαθεστώτα στην Κρυμαία. Και οι Εβραίοι εκεί έχουν αλλάξει στάση και παρουσιάζουν οι ίδιοι κομμουνιστές και αριστεροί και το Ισραήλ ως φασιστική χώρα. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή βγήκε από την κοινότητα ανεξαρτήτων κρατών και φυσικά μετά οδηγήθηκε προς το ΝΑΤΟ ως αποτέλεσμα της προσάρτησης όλα αυτά. Όσο για το σύμφωνο της Βουδαπέστης, πώς θα καθησυχάσουμε τους Ουκρανούς και θα τους ζητήσουμε να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα αν έχουν να αντιμετωπίσουν τις απειλές, τις στρατιωτικές απειλές. Η Ουκρανία είχε πει ότι θα παρατούσε το πυρηνικό της πρόγραμμα εάν είχε εγγυήσεις άλλου είδους. Επίσης με ανησυχεί γιατί μιλήσατε και για την Τουρκία. Η συμπεριφορά του Ερντογάν όντως έχει γίνει περίεργη. Και τελικά η Τουρκία δεν ξέρω αν θα έκλεινε τα στενά των Δαρδανελίων σε περίπτωση επίθεσης του Πούτιν. διότι μετά την προσάρτηση διαπιστώνουμε ότι η Τουρκία τελικά δεν μπορεί να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το αυταρχικό καθεστώς του Πούτιν. Επίσης έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα από την προσάρτηση και πρέπει να συνεχίσουμε να την καταδικάζουμε απολύτως. Η μόνη ευχάριστη εκπληξή είναι ότι σήμερα το πρωί συνάντησα έναν ανώτατο Ουκρανό αξιωματούχο και έλεγε ότι η κινητοποίηση, η στρατιωτική κινητοποίηση που κάνει η Ουκρανία αυτή τη στιγμή κατέληξε στο ότι μπόρεσαν να αυτοαμυνθούν καλύτερα από ό,τι περίμεναν και δεν εξαρτώνται τόσο από το ΝΑΤΟ η Μαριούπολη δεν ε, έπεσε στη Ρωσία. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα πετύχουν τα σχέδια του Πούτιν με το στρατιωτικό διάδρομο εκεί. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας λοιπόν υπήρξαν πολύ πιο θαραλέες από ό,τι λέμε από την επίθεση από τη Ρωσία. Ευχαριστούμε. Θα έρθετε κι εσείς να ακούσετε την ακρόαση για τα πυρηνικά ελπίζω. Ο κύριος Κέλλαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ένας από τους προηγούμενους ομιλητές είπε ότι πρέπει να τα βρούμε με τη Ρωσία γιατί είναι γειτονά μας. Πριν από 8 χρόνια κάποιος είπε ότι ε, θα έπρεπε να τα βρούμε με το ή να τα βρούνε τότε με το Χίτλε γιατί ήταν γείτονα. Ναι, γείτονα η Ρωσία, αλλά όχι ο Πούτιν. Και ο Πούτιν ανακήρυξε τον πόλεμο στη διεθνή τάξη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς καλούμεθα να αντιδράσουμε. Η έκθεση του συναδέλφου Πάσκου είναι επίκαιρη και χρησιμοποιεί και ειλικρινή γλώσσα γιατί το δίλημα που αντιμετωπίζουμε είναι μήπως ε, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις ή μήπως θα έπρεπε να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι η κατάσταση ασφάλειας και η στρατιωτική έχουν αλλάξει και θα το και ακόμα πιο ισχυρά, δηλαδή με την προσάρτηση της Κρυμαίας η Ρωσία προκάλεσε τη διεθνή τάξη πραγμάτων. Η Ρωσία δηλαδή κατ' ουσίαν γκρέμισε την υπάρχουσα διεθνή τάξη με παράπλευρες απώλειες που έχουν σχέση με την ε, λαθρομετανάστευση, με την ε, ενέργεια και την ε, ανείχνευση άλλων ενεργειακών πόρων. Τώρα, όσον αφορά στην Κρυμαία, η Κρυμαία έγινε βάση της Ρωσίας με περισσότερες ε, στρατιωτικές δυνάμεις και αυτό είναι και συμβολικό γιατί μην ξεχνάτε, μετά από κάποιες λίγες μόνο ημέρες έχουμε την 70η επέτειο από τη συνθήκη της Γιάλτας, που τότε καθορίστηκε το μέλλον της Ευρώπης, των χωρών της Βαλτικής και πολλών άλλων κρατών. Έτσι λοιπόν η Κρυμαία σήμερα έχει και ε, συμβολική αξία. Ας πάμε τώρα πάλι στο δίλημά μας. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι το εξής. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την προσάρτηση της Κρυμαίας. Παθητικά, μόνο λεκτικά, δηλαδή θα περιστούμε μόνο σε δηλώσεις ότι ποτέ δεν θα αναγνωρίσουμε την εξέλιξη αυτή. Εντάξει, είναι και αυτό ένα εργαλείο και είμαστε ενωμένοι, αλλά πρέπει να την δράσουμε και πιο ενεργά. Η Ρωσία θα πρέπει επίσης να δεχτεί ε, πιο επιθετικές πολιτικές ε, που θα ξεκινούν από τη Μαριούπολη, από την Οδυσσό ε, σε σχέση με την υπερδνηστερία και συμφωνώ με έναν Ουκρανό σχολιαστή που είπε ότι αν δεν υπήρχαν οι κυρώσεις τότε η Ρωσία θα είχε ήδη προσαρτήσει και την Οδυσσό. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση να διαφυλάξουμε τις κυρώσεις. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πιέσεις, ασκούνται πιέσεις για να χαλαρώσουν οι κυρώσεις. Εμείς δεν τα καταφέρνουμε πολύ καλά ε, και όσον αφορά την υφαλιότητα και επειδή έχουμε διστάσει πάρα πολύ πράγματι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι η Κρυμαία είναι σημαντικό σύμβολο για την πολιτική μας. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να περιμένουμε θετικά μηνύματα από τη Ρωσία, από το γειτονά μας. Όσο η συμπεριφορά της είναι επιθετική και όσο η Ρωσία ανατρέπει τη διεθνή τάξη πραγμάτων, πρέπει και εμείς ε, να αποδίδουμε ε, τα ίσα. Ο κύριος Μπουστινάρο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά που είναι ρεαλιστική, ψύχρεμη προσέγγιση και ρεαλιστική εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα. Και για όσους ε, χάνουν λίγο τη γενική εικόνα αναφερόμενοι μόνο σε λεπτομέρειες, θέλω να σας πω ότι στην ευρωπαϊκή ιστορία το ίδιο λέγαμε κάποια εποχή στο Χίτλερ ή για το Χίτλερ, γιατί λέγαμε ότι ήταν πολύ δυνατός και πρέπει να ζήσουμε μαζί του. Μετά τη συμφωνία του Μονάχου περάσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέπουμε τώρα την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα γενικότερα και στην Κρυμαία ειδικότερα. Πιστεύω ότι η εικόνα και η ρωσική στρατηγική είναι πολύ ευρύτερη και πολύ πιο επικίνδυνη. Πρέπει τη Μαύρη Θάλασσα και την Κρυμαία να τα συσχετήσουμε με την Νότια Οσετή και την Απχαζία. Μην ξεχνάμε τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση μεταξύ Ρωσία και Οσετία που συζητήθηκε στην Επιτροπή μα και θεωρήθηκε τότε μια πολύ επικίνδυνη πτυχή. Δεύτερον, πρέπει να το σκεφτούμε όλο αυτό το θέμα με την υπερθυμιστερία η Ρωσία μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις επομένως σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή. Και δεν είναι μόνο αυτή η γη της ε, Κρυμακής Χερσονήσου που το είπαν και πολλοί άλλοι. Μετά την κατοχή που έγινε κατά του διεθνούς δικαίου, βαρύ στρατιωτικός εξοπλισμός αναπτύσσεται στην περιοχή. Είναι για την πλάκα για λόγους ιστορίας, για να κάνουν στρατιωτική διακοπές στην Κρυμαία που είναι καλές εγκαταστάσεις. Όχι. Είναι τουλάχιστον 35 καταδιοκτικά μαχητικά τζέτα από τα πιο σύγχρονα ε, των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, 1,7 δις εξυγχρονισμός αεροδρομίου και για την υποστήριξη του στόλου του Ρωσικού στην Μαύρη Θάλασσα και 300 πύραυλοι Σκάντερ που μπορούν να αναπτυχθούν και όπως λένε να το εκεί έχει ίσως ανάπτυξη πυρηνικών δυνατοτήτων να αναπτύσσεται στην Κρυμαία από τη Ρωσία. Όλα αυτά τι είναι. είναι. Ένα παιχνίδι με την ιστορία και τα χειρίδια της ιστορίας. Όχι, είναι κάτι παραπάνω. Είναι μια σαφής πρόκληση τα μαχητικά αεροσκάφη της Ρωσίας παραβιάζουν ε, διαρκώς ε, τον εναέριο χώρο και χωρών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και της Τουρκίας. Πολύ παρόμοια η κατάσταση με ό,τι συνέβη στην Μαύρη Θάλασσα. Και έχουμε και μια άλλη διάσταση της ασφάλειας, προμήθεια φυσικού αερίου, που θα έπρεπε να το σχετίσουμε με την ασφάλειά μας. Ο αγωγός South Stream υποτίθεται θα εντασσόταν στην ε, προμήθεια αερίου από τη Ρωσία ε, στην Ευρώπη έχει κολλήσει προς το παρόν. Αλλά μας δημιουργεί μεγαλύτερη εξάρτηση πλέον αυτή η κατάσταση ενεργειακή από την Ρωσία και μεγαλύτερη ευαλωτότητα ε, μας δημιουργεί. Είναι και ένα σημείο της παράθεσης μεταξύ Ευρώπης και ΝΑΤΟ αφενός και Ρωσίας αφετέρου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα Μιστράλ μπορούν με τον πλέον δραματικό και επικίνδυνο τρόπο να αλλάξουν τις ισορροπίες στη Μαύρη Θάλασσα, εάν αυτά τα πολεμικά πλοία κάποια στιγμή αναπτυχθούν. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέατρο επιχείρησεων. Δεν υπήρξε καμία πρόκληση από τον ΝΑΤΟ, από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία που να σα πω και όλε ότι είναι και πλήρη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ολοκληρώνω με μια τελευταία πρόταση. Εάν κάποια μέρα, κοιτώντα από την Ισπανία, αυτέ οι μικρές λεπτομέρειες, Βουλγαρία, Ρουμανία, είναι λιγότερο σημαντικά, σκεφτείτε ότι αυτό το θέμα αφορά όλους μας και τους 28 και όχι τη με την άλλη χώρα. Κάποιες φορές πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας Ευχαριστώ. Thank I would like to, ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω τώρα από τον εισηγητή μας, τον κύριο Πάσκου, να προβεί καταληπτικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ καταρχάς όλες και όλους εσάς για τις παρεμβάσεις σας και για την υποστήριξη αλλά και την κριτική που ασκήσατε. Αυτό περίμενα άλλωστε, γιατί μόλις πήρα αυτήν την έκθεση, αμέσως άρχισα να δέχομαι τηλεφωνήματα από διάφορες πλευρές για το ποια θα είναι η κατεύθυνση της έκθεσης. Υπήρχαν ε, δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες προσδοκίες και όλα αυτά λοιπόν επιβεβαιώνονται σήμερα σε αυτή την πολύ ζωντανή συζήτηση που είχαμε. Θα προσπαθήσω να δώσω σύντομες απαντήσεις σε ορισμένα από τα ερωτήματα και προβλήματα που ετέθησαν. Καταρχάς συμφωνώ με τον κύριο Λαντσμπέργκης. Πρέπει. Σίγουρα να χαράξουμε μια στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα. Η Κρυμαία είναι στη μέση. Είναι η πρόκληση για όλα όσα αναφέραμε. Αλλά ξέρετε, αλλάζει τελείως την εικόνα και το τοπίο. Και ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να είχαν μια περιφερειακή προσέγγιση για αυτή την περιοχή, όπου θα εντασσόντουσαν σε αυτή την προσέγγιση και κάποια μέτρα. Και όλα αυτά θα δημιουργούσαν μια de facto στρατηγική. Μπορεί να μην είχε σχεδιαστεί, αλλά τέλο πάντων θα ήταν εκ των πραγμάτων μια στρατηγική τελικά. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει ένα δόγμα για τη Μαύρη Θάλασσα για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις πτυχές που αναφέρθηκαν με τον κύριο Γιούρεκ, ναι, συμφωνώ αυτό που είπατε για την πολιτική διάσταση του προβλήματος που είναι πολύ σημαντική. Θα σα δώσω δύο παραδείγματα. Για μα, αν θέλουμε να αναθερμάνουμε τη συνεργασία μας με τη Ρωσία, που μακροπρόθεσμα είναι κάτι αναπόφευκτο και αυτό πρέπει να πράξουμε, πρέπει αυτό να το κάνουμε χωρίς να φανεί ότι δεχόμαστε την προσάρτηση. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό όμως, δηλαδή να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα στους Ρώσους, χωρίς να ερμηνευτεί αυτό όμως ως δείγμα δυναμίας από πλευράς μας. Εξίσου, εάν κάνουμε ένα βήμα προς την πλευρά του κυρίου Πούτιν, ο οποίος αύξησε τη δημοτικότητά του, ψώντας το ανάστημά του απέναντι στις κτλ. κτλ. Δεν μπορεί τώρα να δεχθεί κανένα συμφιλιωτικό βήμα γιατί θα το παρερμηνεύσουν οι δικοί του. Ορίστε που είμαστε λοιπόν. Αυτό είναι το πολιτικό τοπίο. Είναι πολύπλοκο. Έτσι έχουν όμως τα πράγματα. Αλλά συμφωνώ ότι πρέπει και τα πολιτικά ζητήματα να μας απασχολήσουν. Γεωργία για παράδειγμα. Την παραγνωρίσαμε εντελώ. Δεν πήραμε τα μηνύματα. Και να τι μας ξημέρωσε. Η Γεωργία όμως, η Απχαζία, η Νότια, η Οσετία, η Ρωσία λέει ξεχάστε τα αυτά, πάνε αυτά στις διεθνείς διασκέψεις το λένε ανοιχτά. Πρέπει αυτά τα προβλήματα να τα δούμε και να τα εντάξουμε στην όλη αυτή, ε, στο όλο αυτό δόγμα μας, αν για τη Μαύρη Θάλασσα. για το Κωσυφοπαίδιο, οι συνάδελφοί μου σας είπαν ότι υπήρξε κίνδυνος γενοκτονίας εκεί. Πρέπει να σταματήσει. Αλλά στην Κρυμαία δεν υπήρχε Κίνδυνο γενοκτονία ούτε για τους ούτε για κανέναν. Και αυτή είναι η διαφορά. Και ο Στάνοκ είπε ότι δεν υπάρχει από ηθική πλευρά καμία σύγκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Τι είχαμε στην Κρυμαία. Είχαμε πράγματι αυτόν υβριδικό πόλεμο. Υπήρχαν αυτοί που όλοι ξέραμε ότι είναι Ρώσοι. Η Ρωσία όμως δεν το δεχόταν ότι είναι Ρώση αυτή Και ανοίγω μια παρένθεση. Θα ήθελε η Ρωσία μια λύση στην κατάσταση για την Ουκρανία. Δεν αναγνωρίζει όμως ότι είναι μέσα σε αυτή τη σύγκρουση, ε, ότι είναι ε, μία από τις πλευρές της αντιπαράθεσης. Άρα επισήμως γιατί να είναι συνομιλητής μας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι συνομιλητής μας, αλλά άμα δεν δέχονται και δεν αναγνωρίζουν ότι είναι μέρος αυτής της σύγκρουσης, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία που θα ήθελαν όμως και οι Ρώσοι να ξεκινήσει. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός λοιπόν ότι ελέγχουν τα στρατουκές. Και έχουμε και την προέλαση των αυτονομιστών προς τη Μαριόπολη και δεν ξέρουμε τι θέλουν να κάνουν τελικά. Αν θέλουν να ελέγξουν εντελώς τη θάλασσα του Αζόφ, που ίσως και να την ελέγχουν ήδη. Η Τουρκία τώρα που ελέγχει το, Βόσφορο, το Βόσπορο και τα Δαρδανέλα. Δεν σημαίνει ότι ελέγχει όμως τη Μαύρη Θάλασσα. Εξ ολοκλήρου. Αν δεχθούμε το επιχείρημα για τα στενά του Κέρτ, θα πούμε ότι η Τουρκία ελέγχει την, ε, το Μαύρη Θάλασσα. Δεν λειτουργούν έτσι αυτά τα πράγματα. Και αυτό το επιχείρημα πρέπει να το ξεπεράσουμε για την υπερθυνιστεριά που δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Δεν έχει σχέση όλο αυτό με αυτό που θέλει να πετύχει η Ρωσία. Η μόνη διαφορά, αν θέλετε, είναι ότι η ιστερία έχει ρωσικά στρατεύματα που είναι ως φιλιρινική δύναμη εκεί, ειρηνευτική δύναμη. Είναι μολδαβική επικράτεια, ενώ η Κρυμαία είναι ρωσική τώρα επικράτεια. Και κάτι άλλο, αυτό ισχύει για το Καλίνιγκραντ που θα πω τώρα, που ανήκει στη Ρωσική επικράτεια. Δεν είναι έτσι κάτι στον αέρα που κάπου αλλού ανήκει και τυχαίνει να έχει εκεί κάποιο στρατεύματα η Ρωσία. Από νομική πλευρά υπάρχει διαφορά. Όμως, κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε, το σχέδιο είναι να έρθει στον έλεγχό του η Οδυσσός. Και όπω και η Ανατολική Ουκρανία, η Οδυσσός τότε θα εντάξει, θα προσαρτήσει την υπερνηστερία. Για διαβάστε κάποιες τοπικέ εφημερίδε από την Οδυσσό και θα τα δείτε όλα εκεί. Μου το έχουν πει οι φοιτητέ μου. Τα γράφουν οι Ρώσοι εφημερίδες. Δεν είναι λόγια του αέρα. Α, μόνο την Ουμανιτέ διαβάστε εσείς, οι άλλες δεν μετράνε, μάλιστα. Ρουμανικός εθνικισμό στη Μολδαβία. Δεν μπορώ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση εδώ. Από τη στιγμή που Πολυδαβή είναι ρωμανικής προέλευσης, ε, γιατί μιλάμε για ρουμανικό εθνικισμό, εντάξει, μπορώ να δεχθώ αυτά που είπατε. Αλλά δεν βλέπω κάποια άλλη σχέση. Η διαφορά μεταξύ Ρωσίας και Ρουμανίας, ξέρετε ποια είναι ότι η Ρωσία την Κρυμαία τη θεωρούσε έδαφος της εδώ και εκατοντάδες χρόνια την κατέλαβαν ακριβώς με το επιχείρημα ότι τους ανήκει, ενώ η Ρουμανία δεν εισέβαλε στη Μολδαβία να την κατακτήσει με το ίδιο επιχείρημα ότι μέχρι το 1811 ανήκε σε αυτήν. Αυτή είναι η διαφορά. Μπορείτε να ολοκληρώνετε, λέει πρόεδρος. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. προσπαθήσω. Να μην πούμε και στην σύμβαση του Μοντρέ, που είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα και λεπτά ζητήματα, να μην μπω σε αυτό, σε αυτά τα χωράφια. Ναι. Όταν υπεγράφει το 1936 συμφωνία του Μοντρέ, δεν υπήρχαν ελικόπτερα. Ο κ. Σικόρσκι έπαιζε ακόμα, ε, πειραματιζόταν με αυτήν την ιδέα. Δεν υπήρχαν ε, ελικόπτερο φόρα. Τέλο πάντων, το όλο θέμα είναι πολύ λεπτό. Για τον άλλο κύριο εκεί, τον κύριο Κόζο. Είπατε ότι είπα θέλει να κρατήσει την Ευρώπη και τη Ρωσία σε αντιπαράθεση. Θα σας πω κάτι που δεν είναι καινούριο, ότι η Ρωσία θέλει να κρατήσει ε, σε αντιπαράθεση μακριά τη, ΣΥΠΑ από την Ευρώπη. Άρα οι μεν κατηγορούν τους δε και οι δε τους μεν. Για τον κύριο Τάραντ. Είναι ο μόνος πράσινος που αναγνωρίζω επειδή είναι πράσινη η κάρτα του. Αστείο ήταν έτσι, μην το πάρετε σοβαρά αυτό που είπα. But, um, I think... Πιστεύω ότι τα επιχείρηματά του όμως ήταν πέραν του αστείου σωστά. Αν βγάλουμε τα κράτη από τον Άτο, τι μένει, τίποτα. Ε, ο κύριο Κέλλαν τώρα έκανε ένα ερώτημα. Πώς θα αντιδράσουμε. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα. Και εδώ είναι και η μεγάλη πρόκληση της όλης έκθεσης. Τι συστάσεις πρέπει να διατυπώσουμε. Πώς πρέπει να αντιδράσει η Δύση και πώς πρέπει να συνεχίσει να αντιδράει η Δύση. Θέλω επίση να αναφέρω ότι θα συμπεριλάβω μνήα και στα ανθρώπινα δικαιώματα παρότι μιλάμε για στρατιωτική περίπτωση, για να, ληφθούν για να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των Ρώσων πριν στην Κρυμαία, αλλά και η κατάσταση των Τατάρων τώρα στην Κρυμαία, γιατί έχει υπάρξει αλλαγή καθεστώτος. Και η παράγραφος, η σχετική, πρέπει να συμπεριληφθεί, πιστεύω, στην έκθεση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση που αφορά στην στρατηγική και στρατιωτική κατάσταση στην Μαύρη Θάλασσα μετά την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας. Η πρώτη συζήτηση επί της έκθεσης ε, θα λάβει χώρα στις 26 Φεβρουαρίου και η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 3η Μαρτίου μέχρι το μεσημέρι. Και τώρα περνάμε πάρα αυτά στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η μαρτιου μεχρι το μεσημερι και τωρα περναμε παρα στο έκθεση για την ε, εφαρμογή της ΕΚΠΑ και εδώ θα ακούσουμε την έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Αυτά για το 2013. Ο κύριος Ντανζόν ε, είναι ο και παρακαλώ έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για τη έκθεση, η οποία εντάσσεται σε ένα διάστημα μεταξύ δύο ε, συμβουλίων που αφορούν την άμυνα Δεκεμβρίου του 2013 και του Ιουνίου του 2015 που επίκειται, αυτές είναι οι προθεσμίες, μπαίνει στο μεσοδιάστημα λοιπόν αυτή η έκθεση και θα επικεντρωθεί στα ζητήματα τα οποία ε, εντόπισε το Συμβούλιο του 2013 και που είναι ένας οδικός χάρτης μέχρι τον Ιούνιο του 2015 που έχουμε το επόμενο Συμβούλιο για θέματα άμυνας. Κάποιοι συνάδελφοι ίσως θα πίστευαν ότι η έκθεση θα είναι πλήρης, διεξοδική, αναλυτική και θα καλύπτει όλες τις αποστολές και επιχειρήσεις της ε, κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Δεν είναι αυτό όμως το θέμα. Αυτό το οποίο προτίμησα να κάνω είναι να αντιγράψω κατά κάποιο τρόπο τον οδικό χάρτη που δόθηκε και στον Οργανισμό Άμυνας το 2013 από το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μορφή της έκθεσης, ε, έχουμε περιορισμό. Δεν μπορεί να είναι 50 σελίδες η έκθεση. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα μέσα. Γι' αυτό και είναι πολύ συνθετική η έκθεση. Μπορείτε να καταθέσετε και τις τροπολογίες σας, αλλά επισημαίνω ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε έναν πλήρη κατάλογο για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε και ένα πολιτικό μήνυμα προς το Συμβούλιο, αλλά και προς την κοινή γνώμη βέβαια. Τρίτο σημείο για τη μορφή πάντα και σχετίζεται με τα δύο προηγούμενα. Δεν δίνω λεπτομέρειες για κάποιες κρίσεις ή κάποιες συγκρούσεις που θα δικαιολογούσαν μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επέμβαση. Και επειδή προκαταλαμβάνω ήδη τις τροπολογίες σας, εννοώ την Ουκρανία. Είναι μια ανοιχτή σύγκρουση ε, στις θύρες της Ευρώπης. Και είναι και σίγουρα ένα θέμα μίζωνος ανησυχίας. Δεν είναι όμως το αντικείμενο αυτής της έκθεσης. Σας υπενθυμίζω ότι σαφώς από την αρχή της Ουκρανικής κρίσης τα κράτη-μέλη δήλωσαν ότι δεν θα δώσει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση Ευρωπαϊκή Ένωση έξω και δεν επιμένω εγώ στην έκθεσή μου σε λεπτομέρειε για το πώ εξελίσσεται η κατάσταση στην Ουκρανία, ούτε και στην εξέλιξη κατάσταση στο Μάλι, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή και στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι αντικείμενο αυτή τη έκθεση. Δεν κάνω απολυσμό όλων των συγκρούσεων για να δω τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθώ να είμαι πιο συνθετικό, πιο περιεκτικό. Σίγουρα με αυτέ τι ε, συγκρούσει ε, ε, στο μυαλό έχω κάνει κάποιες προτάσεις. Τώρα, ποια είναι η διαπίστωση που διέπει την έκθεση. Είναι μια ομή βία η διαπίστωση ότι η Ευρωπαϊκή Ήπειρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως ποτέ από τότε που δημιουργήθηκε δεν περιβαλλόταν σε τόσο μεγάλο βαθμό από απειλές, συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις. Όπου και αν στρέψουμε το βλέμμα μας νότια, δυτικά, ε, νότια, ανατολικά, νοτιοανατολικά υπάρχουν κρίσεις οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ασφαλειά μας. Και με βάση αυτό διαπιστώνουμε ομά ότι ούτε στην περίπτωση της Ουκρανίας, ούτε στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής, ούτε στη Συρία και στο Ιράκ, τη Λιβύη, το Σαχέλ, σε καμία κρίση δεν επιβληθήκαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας πρωταγωνιστής μείζον παίκτη. Στην καλύτερη περίπτωση είμαστε ένα από του εμπλεκόμενου φορεί. Τι περισσότερε φορέ όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση δρά διάχυτα, ε, κατακαιρματισμένα μέσω των κρατών μελών που έχουν διαφορετικέ πολιτικέ και κριτήρια το ένα από το άλλο. Και όταν παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό γίνεται πολύ λίγο, πολύ αργά και με πολύ μικρό συλλογικό τρόπο. Αυτή η διαπίστωση λοιπόν διέπει την έκθεση όπως και το Συμβούλιο του 13 σε ένα βαθμό, που είπε ότι θα πρέπει την πολιτική άμυνα και ασφάλειας να τη θεωρήσουμε προτεραιότητα. Μπαίνουμε τώρα στο ψητό. Ποια είναι τα σημεία του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013. Τι διαπιστώνουμε, δυστυχώς. Απέχουμε πόρο του να έχουμε πετύχει. Είχαμε αναλάβει δεσμεύσεις, είχαμε δηλώσει τις φιλοδοξίες μας που τότε και μετριοπαθείς τις ε, θεωρούσα ένα χρόνο μετά τι διαπιστώνουμε, ότι πόρο απέχουμε το να έχουμε πετύχει κάτι. Πανέρχομαι σε κάποια σημεία. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και τις αποστολές, διαπιστώνουμε και τονίζουμε εκ νέου τα διαρθρωτικά κενά, για μια ακόμη φορά αναφέρθηκε το πρωί και εμβαθύναμε σε αυτό, είναι η χρηματοδότηση, παραμένει κρίσιμο θέμα, ιδίως μεταρρύθμιση, αναθεώρηση του μηχανισμού Αθηνά, Διαρωτώ με. Πάλι μπορεί να το βρείτε λίγο ομό κάποια από εσά. Διαρωτώ με. Πώ οι μη στρατιωτικέ αποστολέ τη Ένωση, τη ΚΠΑ, υποτίθεται ότι είναι και η προστέμενη της τη Ευρωπαϊκή Η καθολική γενική μας προσέγγιση εδώ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους διεθνούς οργανισμούς. Αυτές οι μη στρατιωτικές αποστολές αν τις δει κανείς από πιο κοντά, δεν προσφέρουν αυτή την προσθέμενη αξία. Λόγω προβλημάτων ε, λειτουργίας, δυσλειτουργίας για να είμαι πιο ακριβής και τα υπογραμμίσαμε αυτά τα προβλήματα μεταξύ των διαφόρων οργάνων στις Βρυξέλλες ε, επιτόπου. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των χωρών, ποιες μπορούν να παρέμβουν, να αναπτυχθούν εκεί και τι μπορούν να προσφέρουν και κάποια κενά που υπάρχει υπάρχουν μεταξύ του εύρους της κρίσης και της δικής μας μετροπερθούς προσέγγισης και ανάπτυξης. Έχουμε τη διαχείριση συνόρων στη Λιβύη. Αυτή η αποστολή δεν έχει καμία σχέση με, σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας. Εξού και η πνότη αυτή τη στιγμή. Και δεν έχει εντελώς ακυρωθεί ακόμη και καταργηθεί γιατί θέλουμε να προετοιμάσουμε κάτι καλύτερο στο μέλλον ίσως. Πρέπει να διαρωτηθούμε λοιπόν και να θεωρήσουμε στρατηγικώς τι προσφέρουν οι κάθε από αυτές τις αποστολές επιχειρήσεις και πώς τις αντιαχειριζόμαστε. Στρατιωτικές επιχειρήσεις τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δρά πολύ σε αυτό το επίπεδο γιατί υπάρχουν άλλοι οργανισμοί. Έφυγε ο συνάδελφος που τα λέει καλύτερα από με. Τέλος πάντων. Παραδόξως όμως μάλλον καλύτερα τα πάει ένας με τις αυτιωτικές επιχειρήσεις. Ίσως γιατί, εντάξει, μπορεί να μην γνωρίζουν, να μην έχουν τα ίδια προβλήματα σε ό,τι αφορά τη δίκη και τη διοικητική μέρα με τις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και απ' την άλλη, γιατί σήμερα, με εξαίρεση την Αταλάντη και την Αλτέα, έχουμε εμπειρία, γιατί ε, είμαστε στην, ε, στον τομέα της κατάρτισης, εκπαίδευσης στο Μαλί ε, το έχουμε δει και Σομαλία και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το ίδιο μάλλον θα ισχύει. Έχουμε εμπειρία λοιπόν σε αυτούς τους τομείς. Όμως, η ΕΚΠΑ που είναι πολιτική διαχείριση κρίσεων δεν είναι όμως το train και equip, κατάρτιση εξοπλισμός, δεν είναι αυτός ο πυρήνας αυτής της πολιτικής. Διαχείριση των κρίσεων είναι ο πυρήνα. Άρα εδώ έχουμε ένα στρατηγικό ερωτηματικό για κατάρτιση, εκπαίδευση των ε, ε, ξένων στρατευμάτων θα οργανώσουμε αυτές τις αποστολές. Ναι. Από τη στιγμή που στην προκειμένη περίπτωση θέλουμε διαχείριση κρίσεων περισσότερο. Τα κράτη-μέλη όμως ε, δεν ε, παίρνουν εύκολα το ρίσκο, δεν θέλουν να αναπτύξουν άμεσα δυνάμεις επιτόπου και ούτω καθεξής. Και είναι πολύ λίγα τελικά αυτά τα κράτη που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με εξαίρεση της ε, αποστολής στο Μαλί, όπου συμμετέχουν 23 κράτη-μέλη, στις τέσσερις άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, κάθε μία έχει λιγότερα από έξι μέλη κράτη-μέλη. Αυτά σε ό,τι αφορά τι στρατιωτικές επιχειρήσεις, δυνατότητες, capacities. Και εδώ έχουμε οικονομικά προβλήματα, δύο θα αναφέρω. Η μεγάλη, τεράστια πλειοψηφία των κρατών μελών δεν είναι στρατοικά πρότυπα του 2% αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο του προπολογισμού όπως και αν δούμε τα νούμερα, δεν φτάνουν στο 2%. Και πολλά προβλήματα απορρέουν από αυτό. Δεύτερον, πιο συγκεκριμένο, το Συμβούλιο είπε ότι πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο συγκέντρωσης και από κοινού χρήσης. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που κάνουν στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, όταν αγοράσουν ευρωπαϊκό εξοπλισμό από κοινού, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο ΝΑΤΟ, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμω. Θέλουμε πράγματι να έχουμε μια συγκέντρωση και κοινή χρήση πολύ ακριβού εξοπλισμού, όμω πάλι απέχουμε πάρα πολύ από το να το έχουμε πετύχει αυτό και υπάρχουν εμπλοκέ. Δεν φταίει η Κομισιόν ε, ε, γι' αυτό, αλλά τα κράτη-μέλη, πρωτεύουσε. Πρέπει όμω ε, αυτή την αντίφαση και αυτό το πρόβλημα το αναφέρουμε. Υπάρχει πάντως ε, δυνατότητα συνεργασίας για ευαίσθητο κρίσιμο εξοπλισμό. Αυτό είναι θετικό. Βέβαια, δήλωση προθέσεων είναι προς το παρόν. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι συγκεκριμένο παρά τις προσπάθειες και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Πρέπει να ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν αυτή τη συνεργασία. Βιομηχανικό επίπεδο. Πάντα η ίδια προειδοποίηση προσοχή. Την αμυντική βιομηχανία να μην τη θεωρήσουμε μια κλασική βιομηχανία. Δηλαδή, να μην τη δούμε μόνο μέσω των κανόνων του ανταγωνισμού και της αγοράς. Αν δεν καταλάβουμε ότι οι αμυντικές βιομηχανίες επηρεάζουν πολύ πιο στρατηγικά τα πράγματα και δεν είναι ο στόχος τους ο μόνος ε, να παραγάγουν ε, ένα ε, φασολάκι ή ένα μπουκάλι απορριπαντικού. Έχουμε την αμυντική βιομηχανία που έχει θέσει εργασίας, πάρα πολύ ευαίσθητες τεχνολογίες. Δεν πρέπει να χάσουμε τον έλεγχο, γιατί δεν τον ξαναβρούμε και θα εξαρτηθούμε από άλλους. Όλη η πολιτική άμυνας και ασφάλειας ε, οδηγεί, έχει το στόχο της στρατηγικής αυτονομίας και δεν πρέπει να το φοβόμαστε αυτό, πρέπει να το αναφέρουμε. Δηλαδή να μπορεί η Ένωση να εξασφαλίζει ε, την ασφάλειά της, την άμυνά της, χωρίς να εξαρτάται από κανέναν. Και βέβαια έχουμε και την συμμαχία μας, την Ευρωατλαντική Συμμαχία, που είναι ακρογωνίως λίθος της συλλογική άμυνας. Αυτά σε αδρότατες γραμμές, αυτή είναι η φιλοσοφία της εκθεσής μου και βέβαια είμαι όλος αυτιά για να μου πείτε πώς μπορώ να βελτιώσω περαιτέρω αυτή την έκθεση αλλά να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για να μην γίνει αυτό το έγγραφο ένας πάρα πολύ γενικός κατάλογος και χάσει εντελώς την πολιτική του ουσία. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Ντανζάν. Ο κύριος Σταγίνα Πιτσόλα είναι σκιώδης για τους σοσιαλιστάς αλλά λείπει. Η κυρία Άννα Γκόμες στη θέση του. δικά σχόλια θα κάνω. Εγώ θα τον αντικαθιστούσα υποτίθεται, αλλά δεν πειράζει, ας τα πει η Άννα. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρνό για την έκθεση του, μου φαίνεται εξαιρετική βάση για την περαιτέρω δουλειά μας. Καταλαβαίνω τους περιορισμούς που έχει χώρου αλλά και από τις δικές του και από τις δικές μας τροπολογίες μπορούμε να τα διορθώσουμε. Πρέπει το έγγραφο να έχει κάποιο σθένος. Συμφωνώ με την ανάλυση του ότι βρισκόμαστε σε τώρα πολύ άσκημη στιγμή ως προς τις απειλές για την ασφάλειά μας. και εσωτερικές απειλές. Οι επιθέσεις στη Γαλλία έγιναν από Γάλλους, γεννημένους στη Γαλλία, αναθρεμένους στη Γαλλία και αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι 3.000 νέοι Ευρωπαίοι που πολεμούν στη Συρία και αλλού. Είναι λοιπόν και δικό μας εσωτερικό πρόβλημα και δεν πρόκειται να λυθεί μόνο με μέτρα ασφαλείας. Πρέπει οι κυβερνήσεις μας να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, διότι οι τελευταίες τους πολιτικές όπως και γελίες, γελία οικονομικά μέτρα προώθησαν τις εξελίξεις που τόνισε ο Γάλλος Πρωθυπουργός όταν μίλησε για το ότι μερικές κοινότητες ζουν σε συνθήκες apartheid. Πρέπει να βελτιωθεί η ασφάλειά μας και δεν έχει γίνει αυτό όπως λέει και η έκθεση του Αρνό Ντανζάν. Δεν πρόκειται μόνο για τη χρηματοδότηση της κοινή πολιτικής αλλά επίσης και τα βασικά πράγματα που οι κυβερνήσεις μας γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνουν για πολύ καιρό και δεν τα έχουν κάνει. Είμαι έξαλλη διότι μόλις επέστρεψα από μία επίσκεψη σε κέντρα υποδοχής της Ένωσης και είμαι πράγματι έξαλλη με αυτά που είδα σε πλήρη αντίθεση με όσα λέμε εδώ συχνά από εμπειρογνώμονες, από συντονιστές, από τις κυβερνήσεις μας, από τα μέλη της Επιτροπής μας κτλ. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν βασικό στοιχείο η ανταλλαγή πληροφοριών όλοι γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους που να γνωρίζουν αραβικά για να παρακολουθούν διάφορες πηγές. Αλλά πολύ λίγα πράγματα γίνονται. Ίσως σε μερικές χώρες μέλη γίνονται, αλλά όχι σε όλες, για να αντιμετωπίσουμε τον εσωτερικό αυτό κίνδυνο και που δεν μπορεί να τον λύσει καμία χώρα μόνη της μόνο πανενωσιακός. Εδώ χρειαζόμαστε την Ευρώπη για αυτό το θέμα και δεν έχουμε τίποτα. Ελπίζω λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την εξαιρετική βάση που μας δίνει ο Αρνόνταν Ζαν για να τονίσουμε ακόμη περισσότερο τι πρέπει να γίνει. Ιδιαίτερα ως προς την συλλογή των πληροφοριών. βλέπουμε αυτή τη γελία έκκληση για τα στοιχεία των επιβατών. Δεν είμαι κατά, αλλά αν πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση για τον έλεγχο της τρομοκρατίας. Για ένα ευρωπαϊκό PNR δηλαδή. Αλλά αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι 15 διαφορετικά συστήματα και κανείς δεν ελέγχει τίποτα. Είναι όμως γελίο οι χώρες μέλη και οι κυβερνήσεις μας να μιλάνε για το PNR σαν να είναι μαγική ράβδος για να λύσει τα προβλήματα που εκείνες θα έπρεπε να λύσουν για τη συλλογή πληροφοριών και τη διάδοσή τους και την ανάλυση τους για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Και μετά η σύνδεση με τις αποστολές μας. Μίλησε ο Αρνό για τη Λιβύη είναι κατάφορο παράδειγμα. Από καιρό λέμε ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε τίποτα όταν ξέρουμε ότι στη Λιβύη δεν υπάρχει καμία δομή διασφάλισης της ασφαλείας εκτός από την εθνοφυλακή και την αστυνομία που ξέρουμε ότι αργά ή γρήγορα θα κυριαρχούνταν από εγκληματικά στοιχεία. Νομίζω ότι με το κείμενό σου Αρνό μπορούμε να βασιστούμε στο κείμενό σου ώστε να κάνουμε κάτι όπως στο ψήφισμα για τη Λιβύη που εγκρίναμε την περασμένη εβδομάδα δηλαδή να χρησιμοποιείται η γνώση που συλλέγεται για τη Λιβύη ώστε να δημιουργηθεί μια σωστή αποστολή ΚΠΑΣΑ για τη Λιβύη. Από το 11 και την πτώση του Καντάφη τα ξέρουμε αυτά και Υπάρχουν βέβαια και άλλοι στόχοι και άλλοι οργανισμοί που θα χρειαστεί να συνεργαστούν όπως ο ΙΕ και τα λοιπά, αλλά το ζωτικό θέμα της οικοδόμησης περισσότερης ασφάλειας είναι ζωτικό και, και για μας. Και δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πρόκειται εδώ για ένα παράδειγμα που αποδεικνύει ότι στην εξαιρετική βάση της δουλειάς του Αρνό μπορεί να γραφτεί μια στεναρή έκθεση. Γιατί οι πολίτες μας οι ίδιοι ζητάνε τέτοιο σθένος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία μου. Ο κύριος Μάρκ Γιούρεκ από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η δική μας πολιτική ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών πιστεύει ακράδαντα ότι το βασικό θέμα της ατλαντικής διάστασης αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή άμυνα. Και για αυτό το λόγο τα περισσότερα κράτη έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Νομίζω αυτό είναι ένα καθοριστική σημασία θέμα για όλες τις απόψεις που ισχύουν στον τομέα της ασφάλειας. Γιατί αν επιθυμούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθούμε στον τομέα αυτό, ε, θα πρέπει να μεριμνήσουμε οι απόψεις μας ε, να συμπεριληφθούν ε, σε μία συνθήκη και να ξέρουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των κρατών μας, συμπληρωματικά βέβαια από αυτά που πρέπει να προσφέρει το ΝΑΤΟ. Υπάρχει η, το πολιτικό όπλο, υπάρχει διπλωματία, υπάρχουν οι συνθήκες και θέλω να επαναλάβω όλα αυτά ορίζονται με ακρίβεια και αφορούν ε, στα κράτη και στα κράτη τα οποία ιδρύθηκαν μετά την κατάρρευση της ε, Σοβιετικής Ένωσης. Οφείλουμε λοιπόν να ορίσουμε με απόλυτη σαφήνεια την εξωτερική μας πολιτική. Όλα αυτά σημαίνουν εμείς επιθυμούμε να αποφύγουμε να χρησιμοποιούνται καταραίοντες μηχανισμοί και αν περιοριστούμε μόνο στη διαχείριση των κρίσεων, νομίζω αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τα τεκτενόμενα, όμως ε, στην περίπτωση αυτή σκόπιμα περιορίζουμε τις ε, δυνατότητές μας παρέμβασης και επέμβασης, άρα δηλαδή ε, δεν έχουμε ουσιαστική αμυντική ικανότητα. Και νομίζω ότι θα πρέπει περισσότερο να αντιμετωπίσουμε την περίπλοκη μορφή των πραγμάτων. Κατόπιν, ένα θέμα το οποίο έρχεται και επανέρχεται στις ε, συζητήσεις μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει παρουσιαστεί με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, παρότι δεν συμφωνώ με όλους τους συναντέλφους που μίλησαν, αλλά φάνηκε ότι επιθυμούμε να υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριοποίηση από πλευράς κρατών εφόσον θέλουμε να είναι και αλληλέγγυα μεταξύ τους. Δηλαδή τα κράτη μας να μπορούν ε, με τον ίδιο τρόπο να υπολογίζουν στην αλληλέγγυα στάση ε, των ε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ, αλλά δηλαδή και των Αμερικανών. Ε, και εδώ ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα ε, στις χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μα πρέπει ε, κανείς να μπορεί να υπολογίζει στη βοήθεια κάποιων κρατών. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι χώρες της Βαλτικής δεν μπορούν να θεωρούν ότι η ανεξαρτησία τους εξαρτάται από τους Αμερικανούς. Όχι, τα δικά μας τα κράτη είναι εκείνα που πρέπει να την ε, ορίζουν. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ουσιαστικά αλληλέγγυοι και ένα τέτοιο μήνυμα ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλαμβάνει μόνη τις ευθύνες της, αυτό οδήγησε στα battle groups, ε, στις ε, μονάδες κρούσης. Τώρα βέβαια πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι ε, οι προθέσεις μας συνοδεύονται και από την αμυντική μας ικανότητα ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα πολιτικό εργαλείο. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει κατά τους ε, επόμενους μήνες. Ε, μια μεγάλη δυναμία των battle groups ε, είναι το ότι δεν μπορούν να κινητοποιηθούν γρήγορα. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους μεγάλα ε, οχηματαγωγά. Στην ε, Μεγάλη Βρετανία, αν θέλετε, υπάρχουν κάποια, αλλά όλα αυτά είναι ένα παράδοξο. Μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ρώσους, αν θέλετε, γιατί εκεί υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς. Και η Ουκρανία έχει αυτή την υποδομή και για την ε, κατασκευή αυτών των ε, αεροσκαφών. Αλλά αν θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε σε θέματα ε, παραγωγής και σε αμυντικά θέματα, νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις χώρες εκείνες των οποίων την ανεξαρτησία επιθυμούμε να διατηρήσουμε και πρέπει να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ουκρανία που ήδη χρειάζεται τώρα βοήθεια, χρειάζεται ηλική βοήθεια και θα πρέπει να της δώσουμε τη δυνατότητα να παράγει, να κατασκευάζει αεροσκάφη. Αν έχετε καλοσύνη να τελειώνετε. Τελειώνω, λέει ο κύριος Γιούρεκ. Λοιπόν, δραστηριοποίηση στον τομέα της και το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να εξυπηρετήσει και να υπηρετήσει την πολιτική. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, ε, γιατί ε, αλλιώς θα καθυστερήσουμε. Τώρα, σκιώδης συγητής. Ευχαριστώ πολύ. καταρχήν θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Ντανζάν για την ξεκάθαρη και τίμια έκθεσή του. Θα επαναλάβω τρία από τα κύρια σημεία του. Πρώτον ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από τη διάσκεψη του 2013 δεν κατάφεραν τίποτα συγκεκριμένο για την εφαρμογή της ΚΠΑ και δεύτερον ότι οι περισσότερες στρατιωτικές και μη επιχειρήσεις έχουν δομικές ελλείψεις. Τρίτον, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ένωσης αφορούν έξι χώρες μόνο, άρα δεν υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από τις υπόλοιπες. «22 δηλαδή χώρες δεν ενδιαφέρονται και αυτό είναι απαράδεκτο». Αυτά είναι όλα προειδοποιήσεις και δυστυχώ αυτό ισχύει. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ντανζάν που μας περιέγραψε την αλήθεια. Τι όμως μπορεί να γίνει. Εκκλήσεις όπως εκείνη στο σημείο 20 της έκθεσης που ζητούν από τα κράτη-μέλη μια για πάντα να αφαιρέσουν όλους τους φραγμούς για τον καθορισμό των battle groups δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τα ίδια αυτά τα battle groups αλλά ολόκληρη την κοινή πολιτική. Και η έκκληση αυτή δεν καταφέρνει τίποτα. Το Συμβούλιο έχει επαναλάβει τη δέσμευσή του να ενδυναμώσει την ΚΠΑ στα τελευταία του συμπεράσματα το Νοέμβριο του 2014. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα ότι η ενδυνάμωση της είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί όπως φαίνεται όπως φάνηκε και τη δεκαετία του 90 οπότε για πρώτη φορά καθορίστηκε αυτή η πολιτική. Θέλουμε πράγματι να την ενδυναμώσουμε και μπορούμε. Αν ναι, τότε πρέπει να καταστρώσουμε ένα μακρόπνο σχέδιο και η χρηματοδότηση της πολιτικής δείχνει μέχρι τώρα ότι οι περισσότερες αλλαγές που χρειάζονται θα απαιτούσαν τροποποίηση της συνθήκης, πράγμα το οποίο είναι τεράστιο πολιτικό παρόβλημα. Ευχαριστώ. Μπότιλ Τσαμπάγιος, σκιώδης για τους πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω τον εισηγητή που διαπιστώνει ότι αυξάνεται η αστάθεια και η ανασφάλεια στον κόσμο. Πρέπει να ξαναδούμε επίσης και τη χάρτα του ΟΗΕ. Δεν συμφωνούμε πάντοτε και για τη στρατηγική αυτονομία. Στη συνθήκη της Λισαβόνας γίνεται λόγος για δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και τέτοια. Πράγματα που τα δεχόμαστε όλοι. Αλλά αν δούμε τους αμυντικούς προϋπολογισμούς των χωρών μελών βλέπουμε ότι μειώθηκαν από την κρίση. Εγώ δεν συμμερίζομαι την ανάλυση σας. Άρχισε πολύ νωρίτερα από την κρίση και ο κυριότερος λόγος ήταν ότι η στρατιωτική απειλή θεωρήθηκε λιγότερο σημαντική από ό,τι πριν. Γι' αυτό μειώθηκαν οι αμυντικοί προϋπολογισμοί. Ενδιαφέρεται περισσότερο το κάθε κράτος για την εσωτερική του ασφάλεια, για την αστυνομία, όχι μόνο για την τρομοκρατία. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει απειλή και αποθεομηνίες. Κρίσεις λοιπόν αντιμετώπιση κρίσεων. Η αστυνομία παίρνει μεγαλύτερη θέση στον προπολογισμό και στρατός λιγότερη. Δεν συμμερίζομαι λοιπόν την ανάλυση σας. Ούτε την άποψή σας να αυξηθούν οι αμυντικοί προϋπολογισμοί. Αυτό που χρειάζεται αντίθετα είναι συνεργασία. Η αγορά της άμυνας είναι πολύ κατακαιρματισμένη και πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Επίσης χρειάζεται μια σωστή ανάλυση του κόστους όλων αυτών. Υπάρχει μια πρόταση για τα ντρόν. Κάποιο νομικό πλαίσιο που να καθορίζει πώς μπορούν και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται. Eh, το Φεβρουάριο του 2014 πριν εκλεγώ φαίνεται ότι είχε τεθεί το θέμα και θα μπορούσε να ξανατεθεί και τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Νάρντ πολύ σύντομα όμως, πάρα πολύ σύντομα σας παρακαλώ κύριε μου γιατί μετά και ο εισηγητής θα απαντήσει σε όλα όσα άκουσε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ντάζαν για αυτό αυτό, αυτό που είπε ότι θα πρέπει να αναλαμβάνουμε όλο και περισσότερο ε, τη δική μας άμυνα. Υπάρχει πράγματι μετατόπιση των ενδιαφερόντων των ΗΠΑ προς τον άξονα Ασίας και όχι στην Ευρώπη. Και επίσης να μην έχουμε μια διμερή διαδικασία ή ε, την ε, ευνοχιστική διαδικασία του μηχανισμού Αθηνά και για την κριτική των Αποστολών Λιβύης και Ράφα και Νέστορ συμφωνώ. Ή να σταματήσουν ή να παγώνουν οι αποστολές ε, εάν δεν ε, δεν έχουν κάποιο, κάποια επιχειρησιακή σκοπιμότητα ή ε, δεν είναι οικονομικά σωστή. Πραγματικά μπορεί να σηκωθούν τα μαλλιά μας ε, άμα δούμε τι δεν συνεισφέρει, πόσο δεν συνεισφέρει σε τίποτα μια εκπαιδευτική αποστολή. Στην υποσαχάρια Αφρική μάλιστα οι εκπαιδευθέντες στρατιώτες είναι καταδικασμένοι να πεθάνουν. Και ολοκληρώνω με τις μάχημες ομάδες, τις ε, τακτικές αυτές ομάδες Σίγουρα όταν υπάρχει πρόκληση θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσονται άμεσα για να δώσουν απάντηση. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την έκθεσή σας. Thank you. Mr. Donjon, floor yours. Κύριε Ντάνζο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Με ενθαρρύνουν και νομίζω ότι έχουμε μία βάση εργασίας πάνω στην οποία θα μπορέσουμε να βασιστούμε για να εμπλουτίσουμε το κείμενο ώστε να ανταποκρίνεται στη γενική κατεύθυνση και προσανατολισμό των πολιτικών ομάδων. Σημειώνω κάτι που είπατε και η Άννα το είπε αλλά και ο Τόνι Πιτσούλα από την ομάδα των σοσιαλδημοκρατών που μου έδωσε ένα χαρτί να ενισχύσουμε αυτή την ε, τη συνέχεια εσωτερική εξωτερική ασφάλεια. Ξέρουμε βέβαια ποια είναι η συγκυρία. Αυτό το συγκρατώ λοιπόν σε ό,τι αφορά τον ΝΑΤΟ. Δύο απλά σχόλια. Πρώτον, δεν έχει νόημα σε κάθε έκθεση να μιλάμε στη σχέση μας και τη διάσπασή μας με τον ΝΑΤΟ. Αυτό το λέει ξεκάθαρα η συνθήκη που αναγνωρίζει χωρίς καμία αφησιμία ότι το ΝΑΤΟ είναι ο ακρογωνίος λίθος της συλλογική άμυνας. Για μένα όμως, ε, για μένα λοιπόν είναι άχρηστο. Μπορούμε να το ξαναλέμε, αλλά γιατί να χαλάμε ε, μελάνι και να λέμε σε παραγράφους συνέχεια τα ίδια για το ΝΑΤΟ. Δεν θέλουμε να αποφύγουμε τον ΝΑΤΟ βέβαια σε καμία περίπτωση, απλά όλα αυτά είναι τα λέει η συνθήκη ξεκάθαρα. Και γιατί να τα ξανασυζητάμε. Δεύτερο θέμα, για τη διάρθρωση και πα ΝΑΤΟ. Το ΙΣΙΑΡ ξέρω ότι πάγια στάση έχει και επιθετική, εγώ ανήκω σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που βρίσκεται και στις ρίζες της δημιουργίας αυτών των αποστολών και πά, υπάρχουν πράγματα που το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να κάνει και σε στρατιωτικό επίπεδο. Δεν μπορεί να πάει παντού, ούτε και με στράτο το ΝΑΤΟ. Η μη στρατιωτική επιχείρηση του Ένωση στη Γεωργία, μόνο από την Ένωση μπορούσε να γίνει. Κανένας άλλος δεν μπορούσε να πάει. Το ΝΑΤΟ ούτε καν, αλλά ούτε και ο ΙΕ, ούτε και ο ΟΑΣΕ. Έχουμε και προβλήματα τώρα στη Βόρεια Αφρική, προβλήματα ασφάλειας. Για ζητήστε από τους Αφρικανικούς ηγέτες, Αφρικανούς ηγέτες και τον πληθυσμό των χωρών εκεί. Θέλουν το ΝΑΤΟ. Να δείτε τι θα σας απαντήσω. Δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να τα κάνει όλα, ούτε και μπορεί να τα κάνει όλα και θέλει να τα κάνει, ούτε και θέλει. Είναι, επαναλαμβάνω, ακρογωνίες της συλλογικής άμυνας και της εδαφικής ασφάλειας, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει χώρος, ίσως περιθωριακά, αλλά υπάρχει χώρος για ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και στο στρατιωτικό επίπεδο. Και αυτό θα το κάνει και η πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Και είναι πράγματι πρέπει να εκμεταλλευτούν ε, την προσθέμενη αξία. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες στις παρατηρήσεις του κυρίου Γιούρικ. ούτε της κυρίας Ερμπάλος. Δεν θα πω αναλυτικά ποιες είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τις δράσεις της ΚΠΑ, δηλαδή σεβασμός εδαφικής κυριαρχίας, κυριότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά είναι γενικές αρχές των δράσεων της ε, ΚΠΑ και περιλαμβάνονται στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, στην ΚΕΠΑ. Εμείς είμαστε μια υποομάδα, αν θέλετε, άμυνας της, ε, της ΚΕΠΑ δεν θεώρησα σκόπα να αναφέρω όλες αυτές τις βασικές αρχές. Γενικά, αν θέλετε, μπορώ να τις επικαλυστώ. Δεν έχω πρόβλημα. Για τη στρατηγική αυτονομία, σε κάθε τη σχέση ε, έκθεση γίνεται αυτή η συζήτηση. Σε ένας προκατόχου σας, τον κύριο Πιτικόφερ, είχαμε μια πολύ τεταμένη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η στρατηγική αυτονομία για μένα δεν είναι μόνο, πώς να το πω, για να είμαστε υπερήφανοι και από κεντρικά να πούμε ότι να ορίστε ποιοι είμαστε στο διεθνές προσκήνιο. Το θέμα να μπορούμε να λέμε και όχι. Παραδείγματο χάρη, κοινή καταστροφική περιπέτεια του 2004 στο Ιράκ, του Αμερικανού φίλου. Στρατηγική αυτονομία θα σημαίνει ότι θα μπορούμε να λέμε όχι. Όταν άλλε χώρε με τι οποίε έχουμε μια κοινή συμμαχία θέλουν να μα παρασύρουν σε περιπέτειες δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Αυτό είναι και η στρατηγική αυτονόμη μεταξύ άλλων. Θέλω να τη βλέπω θετικά δηλαδή. Δηλαδή ότι στην Ευρώπη θα μπορούμε να αναλάβουμε κάποια καθήκοντα που έχουν να κάνουν με τη δική μας ασφάλεια και αν. Διακόπτει ο πρόεδρος. Συγγνώμη κύριε Νταζόν, αλλά θα φύγουν οι διερμηνείς. Τότε να το πω αγγλικά. Τα υπόλοιπα λέει ο κύριος Ντάζο. Ε, θέλω να δουλέψω. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλω να εργαστώ. Δεν θα πεθάνουμε με 10 λεπτά καθυστέρηση. Εμείς θα πεθάνουμε. Να πω στον κύριο Νάτο ότι συμφωνώ με την παρέμβασή του. This afternoon, and I will take a great interest in listening to you, because anyway, I have my doubts about the, the I would say the, the